για τη διαδικασία αυτή. Έχουμε τώρα την εξέταση της έκθεσης Γκερέιδο. Κοινή αλληλευτική πολιτική και προσέγγιση στη χείριση της αλληλείας με βάση το οικοσύστημα. Ο κύριος Γκερέιδο έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η ανακοίνωση βασίζεται, έχει στόχο το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει την εξέλιξη και αλλαγή της κοινή ελευθερικής πολιτικής μετά το 2010. Η έκθεση αυτή ε, παρουσιάζει μια σειρά θεμάτων που θεωρούμε σημαντικά. Η αλληλεία είναι θεμελιώδης δραστηριότητα για την εγγύηση της ίδιας και της επιβίωσης του ανθρώπου, γεγονός που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο κάθε αλλιευτική πολιτική. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία τη αλληλείας στα ύδατα τη αποκλειστική οικονομική ζώνη κάθε κράτου μέρου και την, για την κυριαρχία και εξαντλησία του ιδίω σε επιστημιστικό επίπεδο. Η αλληλευτική πολιτική πρέπει να δίνει προτεραιότητα στα αλληλεύματα και στην βιώσιμη ανάπτυξη τη αλληλείας εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητα σε κοινωνικονομικό επίπεδο και την διαφύλαξη των αλλιευτικών πόρων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να δουν πώ μπορεί να υπάρχει αλευτική ε, ε, ε, επιστημιστική ασφάλεια και βελτιώνοντα το επίπεδο ζωή των εργαζομένων ε, στον τομέα τη αλληλείας. Λαμβάνοντα υπόψη του στόχου αυτού, μια κοινή πολιτική αλληλείας δεν πρέπει να εξαρτάται από άλλε κοινοτικέ πολιτικέ. Δηλαδή, μια αλληλευτική πολιτική δεν μπορεί να είναι μια πολιτική για του ωκεανού ή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Πρώτος στόχος τη διαχείρισης της ω ως δραστηριότητα που εκμεταλλεύεται ένα πόρο είναι ο έλεγχος της ελευτικής προσπάθειας για να εξασφαλίσουμε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αλίευσης. Μια αλιευτική πολιτική πρέπει να ξεκινά από την αλεξάρτηση των αλιευτικών κοινοτήτων και της δυνατότητας να είναι βιώσιμα τα οικοσυστήματα στα οποία μετέχουν, ε, στα οποία εμπλέκονται, αναγνωρίζοντας τον ειδικό χαρακτήρα της μικρής παράκτειας και της παραδοσιακής αλίας. Η εφαρμογή μιας διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με δίκιο τρόπο απαιτεί να να έχουμε μια πολυεπιστημονική και ιδιωτομερική προσέγγιση των πολιτικών που θα είναι άσχετη, ε, που δεν θα είναι κατά ανάγκη αυτοί που υιοθετούνται σε άλλους τομείς αλληλείας, ε, πέραν των ε, άλλων προηλημένων ιδεών, η ανάλυση των αλλιευτικών πόρων πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, ενώ πρέπει να αναγνωρίζουμε ε, τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ρευτικών ζωνών και των πόρων που βρίσκονται στι περιοχέ αυτέ, μεταξύ των διαφορετικών στόλων και τη αντοχή αντοχής των οικοσυστημάτων. Τούτο απαιτεί να υπάρξουν μια σειρά συγκεκριμένων ειδικών και κατάλληλων μέτρων ανά περίπτωση, αντισταθμίζοντας αν χρειαστεί ε, τις συνέπειες ε, που υφίστανται ή αλίες. Για να εξασφαλίσουμε αυτό το κόστος είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να ασκούν την κυριαρχία τους στα 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων που ανταποκρίνεται και στις περιοχές που ανταποκρίνονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των υπερπόντιων εδαφών και που αντιστοιχούν στους δικούς τους πόρους, χρησιμοποιώντας προσφέροντας ένα ειδικό μεταφερόμενο ποσοστό τάκ ανά περιοχή. Είναι σημαντικό ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι δεν δικαιολογείται μια πολιτική η οποία θα ενισχύει την ε, πάυση λειτουργίας κάποιων σκαφών χωρίς ε, να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της διακοπής λειτουργίας τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι αλευτικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να στηρίζονται και μόνο σε στην μείωση των αλευτικών, ότι η, ζωή των αλλιών δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη μείωση των αλευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και στην τιμή του προϊόντος. Η κυρία Βασιλείου έχει το λόγο χαιρετίζει την έκθεση αυτή και την προσέγγιση που σέβεται τα οικοσυστήματα. Ένα, ε, στην ανακοίνωση της η Κομισιόν λέει ότι πράγματι η αλληλεία βασίζεται, εξαρτάται από υγιή οικοσυστήματα. Ωστόσο, η διαχείριση της αλίας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε αυτό. Τα υγεία οικοσυστήματα μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν όλοι οι παράγοντες που πειράζουν τα οικοσυστήματα αυτά είναι ελέγξιμοι. Και η υπάρχει η οδηγία της η, ε, η, οδηγία Marine Strategy που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το περιβάλλον και γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι όχι μόνο η αλία αλλά όλοι οι τομείς οι οποίοι μπορεί να εξαρτώνται από αυτή τη θαλάσσια στρατηγική ε, πρέπει να προστατευθούν ή να βοηθηθούν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μια πολιτική έχει δευτερεύον αθέσεις σε σχέση με κάποια άλλη ότι υπάρχει ιεράρχης πολιτικών στους διάφορους ε, ε, τομείς. Όχι, όταν μιλώ για την οδηγία της ε, θαλάσσιας στρατηγικής εννοώ ότι η οδηγία αυτό έχει την καλύτερη από την πολιτική της Αλίας και τις σχετικές ε, οδηγίες και κανονισμούς αλλά ότι βοηθάει την ε, Γαλλία γιατί ορίζει ε, μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν για να εξασφαλιστεί η υγεία των οικοσυστημάτων που είναι απαραίτητη για την αλληλεία. Ή θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων αυτών συγχρόνως να διατηρηθεί η βιωσιμότητα της ελευτικής δραστηριότητας της, των αλλιέων. Αυτά δεν είναι ασυμβίβαστα πράγματα και η προσπάθεια εξισερώπησης των μεν συμφερόντων με τα δε είναι η πρόκληση για όλους μας για το μέλλον. Δεν θα ήθελα για επειδή βλέπω έτσι τα πράγματα δεν θα ήθελα να απαντήσω συγκεκριμένα σε κάποια ερωτήματα που σχετίζονται με την κοινή αλληλευτική πολιτική ε, αλλά θα ήθελα να δω το θέμα γενικότερα. Αναφέρεται παραδείγματο χάρη ότι κάποιοι αλλοί οι οποίοι επηρεάζονται αν θέλετε από κακά οικοσυστήματα και τα λοιπά θα πρέπει να επιδοτούνται. Όχι, εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε τον κάθε ένα ο οποίος φύσταται μια κάποια ζημία γιατί συνέβη κάτι τι. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τον οικονομικό αυτό κλάδο συνολικά να σταθεί στα πόδια του και να είναι η υδροκαλλιέργεια η οποία αμφισβητείται από ορισμένου ε, επειδή επιδεωτείται σε κάποιο βαθμό και ζητείται να επιδοτηθεί περαιτέρω. Όχι, νομίζω ότι εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε να εξασφαλίσουμε τα λιευτικά αποθέματα να διατηρηθούν σε υγιή κατάσταση για να μπορεί από εκεί και πέρα να δράσει ε, ο αλευτικός κλάδος σωστά το μέλλον θα οργανώσουμε βεβαίως ε, και άλλες συζητήσεις μέσα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα ξεκινήσουμε την πράσινη βίβλο μας τον Απρίλιο και θα γίνουν σχετικές συζητήσεις αργότερα. Προς το παρόν παραμένω εδώ. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε στην τελευταία έκθεση, συνάδελφοι, για την ε, εφαρμογή της ε, Οδηγίας 2273 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανθρώπων και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και την πρόθεση και τις συνθήκες εργασίας. Έκθεση που είναι υπέρ